Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, καθίστε. Έχουμε κάποια καθυστέρηση. Θα είναι σύντομη η συνεδρίασή μα σήμερα, τροποποιημένη σε σχέση με την αρχική ημερήσια διάταξη. Επρόκειτο να μιλήσουμε για διάστημα με τον κύριο Λορέντσιτ, που είναι διευθυντή του κέντρου δορυφόρο του Τορεχών αλλά δυστυχώς ε, είναι ασθενής σήμερα αλλά θα συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με το διάστημα πολύ σημαντικό θέμα και ίσως ε, λιγάκι να παραμελείτε στις εργασίες μας ενώ είναι στρατηγική σημασία ευχαριστώ ιδιαίτερα και ειλικρινά τους ε, ομιλητές μας που μπόρεσαν να έρθουν τόσο σύντομα για να μας μιλήσουν για το σύστημα επιτήρησης του διαστήματος. Ίσως να μην το γνωρίζετε όλοι. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση για αυτό το σημαντικό θέμα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στη συνεδρίασή μας σήμερα, ναι μεν, είναι σύντομη, είναι πέμπτη, μεσημεράκι, έχει μεγάλη σημασία για την υποεπιτροπή μας, διότι είναι η τελευταία συνεδρίαση όπου θα, συμμετά... συμμετέχει ο κύριος Φρανζουλιά, εδώ δίπλα μου, που δεν κάθεται απλώς ε, δίπλα μου, είναι πυλώνας της ε, υποεπιτροπής ως γραμματέας. Λίγη φέτος ε, τέλος της χρονιάς η σταδιοδρομία του. Θα ήθελα να αποτίσω ιδιαίτερο φόρο τιμή στην εργασία του. Η εργασία αυτή είναι συχνά αχάριστη, συχνά γίνεται στα παρασκήνια, αλλά είναι απαραίτητη και δεν θα μπορούσε να είναι γνωστή και η εργασία μας χωρίς αυτόν σε έναν τομέα τόσο ειδικό όπως είναι η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας. Θέλω λοιπόν να τον ευχαριστήσω τον αρμό για την εργασία του με πολύ μεγάλη ευσυνειδησία, αυτό είναι λογικό θα έλεγα, φυσιολογικό, αλλά και με πολύ αποφασιστικότητα. Είναι δύσκολος τομέας η άμυνα, και αυτό φαίνεται και από το καθεστώς μας ότι είμαστε υποεπιτροπή αλλά νομίζω ότι με πολύ προσωπική δέσμευση και αφοσίωση υποστήριξε όχι μόνο την εργασία της υποεπιτροπή μας αλλά γενικότερα την πολιτική, την φιλοσοφία για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και είμαι βεβαίως ότι, βέβαιος ότι και μετά την αποχώρησή του θα συνεχίσει να εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση. Σας παρακαλώ να τον ευχαριστήσουμε. Θα σας επιτρέψω ε, να του δώσω το λόγο στο τέλος της συνεδρίασης για να πει μερικά λόγια ως κλείσιμο πριν ε, αποχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, εισαγωγή. Σας παρουσιάζω τους ομιλητές μας σήμερα. Ο Μάρκο Μαλακάρνε, εδώ αριστερά μου, είναι στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας ε, διευθυντής για τις βιομηχανίες του διαστήματος, την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και την άμυνα. Και η κυρία, θα έπρεπε να έχω ξεκινήσει με την κυρία βεβαίως, συγγνώμη, την κυρία Έλενα Γκρίφωνη Winters της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Διάστημα και ο κύριος Άσμπεκ. Το γνωρίζουμε βεβαίως. στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αρμόδιος σύμβουλος για την πολιτική διαστήματος και την πλευρά της ασφάλειας, κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Το πρόγραμμα αυτό επιτήρησης ε, της κατάστασης του διαστήματος ε, ξεκίνησε το 2009 είναι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα φιλόδοξο που δεν σχετίζεται άμεσα και κατά ανάγκη με τις εργασίες της υποεπιτροπής μας στον τομέα της άμυνας, αλλά έχει πολύ να κάνει με τον τομέα της ασφάλειας. Διότι επιδιώκουμε να αποκτήσουμε την ε, ανεξαρτησία μας για την ε, προστασία των υποδομών που σχετίζονται με την πολιτική του διαστήματος, είτε στο έδαφος είτε στο διάστημα, τους δορυφόρους μας δηλαδή, Υπάρχει μία ολόκληρη προβληματική αντιμετώπιση των θραυσμάτων, των ε, διαστημικών σκουπιδιών. Είναι ένα, πρόγραμμα που, ένα πρόβλημα το οποίο αποκτά όλο και ευρύτερες διαστάσεις, μια που όλο και περισσότερες χώρες ε, ξεκινούν πολιτική διαστήματος και υπάρχει και μία πλευρά άμυνας και ασφάλειας, η προσπάθεια δηλαδή να αντιμετωπίσουμε εχθρικές ενέργειες που μπορεί να γίνουν στο διάστημα κατά των υποδομών μας. Είναι λοιπόν πολύ ευρύ το θέμα. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τους λόγους ύπαρξης του προγράμματος, ε, τον τρόπο λειτουργίας, τις δυνατότητες που έχει συγκεκριμένα, διότι συμμετέχουν ε, αρκετά λίγα κράτη-μέλη και φυσικά τα θέματα χρηματοδότησης και διοίκησης και αυτά είναι πολύ σημαντικά Αυτά θα θέλαμε να μας παρουσιάσει ο κύριος Μαλακάρνε από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νταλζό. Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η παρουσίαση Προ την Επιτροπή σα για να σα εξηγήσω, όπω είπε ο κ. Ντανζό, την λόγους ε, των επεμβάσεων που βλέπει η Κομισιόν σε αυτέ τι περιπτώσει. Μιλάμε για Space Situation Awareness, δηλαδή την επιτήρηση του διαστήματο. Το πεδίο είναι ιδιαίτερα ευρύ. Περιλαμβάνει και αυτό που λέμε για το Space Weather. Και θα ήθελα να εστιάζω στα όσα μόλις ανέφερε ο κύριος Ντανζό δηλαδή το ζήτημα των θραυσμάτων του διαστήματος, τα space junk, σκουπίδια του διαστήματος. Υπάρχουν εκατοντάδες ε, δισεκατομμύρια και έχουν διαστάσεις ε, μερικών χιλιοστών όσο και πολύ μεγαλύτερες. Ε, είναι δύσκολο η κοινή γνώμη να κατανοήσει τι σημαίνει να έχουμε 100-150 χιλιάδες στοιχεία στο διάστημα, αλλά εντάξει και το διάστημα είναι μεγάλο, που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από την γη. Από το, γη. το πρόβλημα όμως ε, γίνεται οξύ στις ε, χαμηλές ε, τροχές, όταν, εκεί που υπάρχουν οι δορυφόροι παρατήρησης. Πρέπει να δούμε τι οικονομική επίπτωση έχει αυτό το πρόβλημα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Όπως ε, ακούσατε, διαβάσατε μάλλον και στις εφημερίδες, ε, οι δορυφόροι χρειάζεται να μετακινηθούν για να αποφευθούν συγκρούσεις. Αυτό συνέβη και πριν από μερικές εβδομάδες ε, στον Διεθνή Σταθμό. Κάθε φορά που ένας δορυφόρος πρέπει να μετακινηθεί από την τροχιά του, καταναλώνει ένα τμήμα του καυσίμου. Το καύσιμο δεν είναι ατέλειωτο και έτσι περιορίζεται ε, η ζωή του δορυφόρου. Αυτό έχει οικονομικές επιπτώσεις ε, που οφείλονται στη μικρότερη διάρκεια ζωής, ε, μέσω όρο διάρκεια ζωής για τους ευρωπαϊκούς δορυφόρους Μιλάμε για 150 έως 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό είναι, αυτός είναι ο οικονομικός αντίκτυπος λοιπόν. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ενδράσει σε αυτόν τον τομέα, αυτό είναι πλούστατο διότι η Ευρώπη είτε σε δημόσιο επίπεδο είτε σε ιδιωτικό διαθέτει με υψηλό αριθμό δορυφόρων, επικοινωνιών, εμπορικού χαρακτήρα, ναυσιπλοείας, πλοήγης κλπ. Και όπως γνωρίζετε εντός ολίγου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει 30 ε, δορυφορικούς και θα είναι άμεση ε, ιδιοκτήτης. Και μιλάω για το Γκάλιλαίο και για το μελλοντικό GMS. Εδώ λοιπόν υπάρχει άμεση ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συντομία, τι προσπαθούμε να πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα αυτών των ε, space debris, των ε, ε, σκουπιδιών διαστήματος. Υπάρχουν τρεις δυνατές λύσεις. Πρώτα απ' όλα αυτή της κατανόηση του πού βρίσκονται αυτά τα αντικείμενα τα οποία είναι δυνάμει επικίνδυνα να τα επιτηρούμε λοιπόν Space Surveillance and Tracking στα αγγλικά και θα πω μερικά λόγια αλλά για να ολοκληρώσω τον κατάλογο των δράσεων υπάρχει ε, κώδικας συμπεριφοράς σε διεθνές επίπεδο και νομίζω ότι σε αυτό γι' αυτό θα μιλήσω ο συνάδελφος Φρανκ Άσμπεκ, ότι αυτή η διπλωματική πρωτοβουλία βρίσκεται υπό την ευθύνη της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν και τεχνολογικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο την εξέβρεση τεχνολογιών που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση και εδώ φαντάζομαι πως η συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ε, που είναι και αρμόδια θα μας μιλήσει για τις ε, τεχνολογικές καινοτομίες ίσως και λίγο φουτουριστικές που προλέπονται για τα προσοχή έτη. Να ολοκληρώσουμε μιλώντας για την δράση του Space Surveillance and Tracking. Αυτό σημαίνει με λίγα λόγια ε, χρησιμοποίηση των μεγάλων ραντάρ, το οποίο βρίσκονται επίγειων ραντάρ, τα οποία ε, προσπαθούν να εντοπίσουν αυτά τα αντικείμενα και ε, προσπαθούν να καθορίσουν την, την πορεία, την τροχιά. Δυστυχώς τα πολύ μικρά αντικείμενα, τα οποία είναι επικίνδυνα και αυτά, ταξιδεύουν με ταχύτητα μερικών χιλιάδων χιλιόμετρων ανά ώρα και οι δυνατότητες επιτήρησης αφορούν αντικείμενα από μεγέθους από μερικά χιλιοστό έως μερικές εκατοντάδες μέτρων. Λοιπόν, και έτσι μπορούμε να έχουμε μία εικόνα γενικότερη. Σήμερα η μοναδική χώρα που έχει ένα σύστημα επιτήρησης των space debris είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη εξαρτάται απόλυτα από τις προφορίες που μας ε, παρέχουν οι συνάδελφοί μας από τις ΗΠΑ, οι οποίοι και αυτοί έχουν κάθε όφελος να αποφύγουν τις συγκρούσεις των αντικειμένων αυτών, διότι μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιες ε, ε, αλυσοειδείς επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή ε, η Κομισιόν προσπαθεί να διευκολύνει τον συντονισμό μέσω ε, μερικών κρατών όπως Γερμανία, Γαλλία και ε, το Ηνωμένο Βασίλειο για την χρήση κατάλληλων ραντάρ που θα μπορούσαν να παρέχουν αν συντονιστούν σωστά σε μια συνεισφορά σημαντική σε αυτό το σύστημα υποκτήρας που καθοδηγούν οι Αμερικανοί. Θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για υποδομές ε, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό τον έλεγχο ε, των στρατιωτικών οντοτήτων, δηλαδή πρόκειται για πρώτη φορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κομισιόν να χρηματοδοτήσουμε άμεσα υποδομές οι οποίες βρίσκονται υπό στρατιωτικό έλεγχο. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κομισιόν θέλουν να επισέλθουν σε ζητήματα στρατιωτικής φύσης, αλλά να μπορέσουμε να λαμβάνουμε πληροφορίες για ε, μη στρατιωτική χρήση, δηλαδή την επιτήρηση των δορυφόρων για μη στρατιωτική χρήση. Πρέπει λοιπόν να συντονιστούν οι διάφορες ε, δραστηριότητε σε εθνικό επίπεδο για να δημιουργήσουμε ένα front desk το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως διαπαθή ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο και τις ε, πολιτικές, μη στρατιωτικές αρχές που ασχολούνται με την διαχείριση των μη στρατιωτικών ε, δορυφόρων. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε προκαταρκτικό διάλογο με τις χώρες που προανέφερα και τις σχετικές ε, εθνικές αρχές. Ελπίζουμε τους προσεχείς μήνες ε, ένα ή δύο χρόνια να καταλήξουμε σε κάποια συνεννόηση, σε κάποια συμφωνία και εδώ σταματήσω για να δώσω το λόγο στους συνάδελφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκριφόνη Βίντερς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, Διαστήματος που οπωσδήποτε συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Θα μιλήσω αγγλικά. Ε, θα συμπληρώσω αυτά που είπε ο κύριος ε, Μαλακάρνε. Ναι. Για ποιο λόγο συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα και ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν την κατάσταση του καιρού στο διάστημα. Πάμε λίγο πίσω για να δούμε τι εννοούμε. Επιτήρηση του διαστήματος. Δηλαδή, να προστατεύσουμε τις υποδομές στο έδαφος και στο διάστημα από απειλές που προέρχονται από το διάστημα. Βεβαίως, αυτά τα διαστημικά σκουπίδια που τα έχει προκαλέσει ο άνθρωπος και κινούνται σε τροχιά, παλιοί δορυφόροι, διάφορα ε, επίπεδα πυράβλων τμήματα διαστημικών σκαφών, διαστημοπλοίων, φακοί τηλεσκοπίων, σταγόνες ψυχτικών υγρών, διάφορα λοιπόν ανθρώπινης προέλευσης αντικείμενα που κινούνται στο διάστημα. Υπάρχει μια ταξινόμηση που περιέχει περίπου 10.000 αντικείμενα Αλλά αυτή η ταξινόμηση, ο κατάλογο τα περιέχει όλα δηλαδή και είναι 10.000, είναι μόνο ε, το 5% αυτών που θεωρούμε ότι υπάρχουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το ESA. Υπάρχουν περίπου χίλιοι δορυφόροι ανθρώπινης προέλευση που κυκλοφορούν γύρω από την γη. Εμείς ελέγχουμε 17 εξ αυτών και σύντομα θα εκτοξεύσουμε άλλου 12. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να του προστατεύσουμε. Ένα άλλο στοιχείο, πολύ σημαντικό για μας, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα των διεθνών διαστημικών σταθμών με άλλους, Ρωσία, Ηνωμένε Πολιτείε, Ιαπωνία. Και οι κοσμοναύτες μας σε αυτούς τους σταθμούς κινδυνεύουν από αυτά τα θράψματα. Το 2012 για παράδειγμα υπήρξαν 50 επίγουσες περιπτώσεις λόγω προσέγγισης τραυσμάτων και κάποιες φορές χρειάζεται να κάνουμε ε, ελιγμούς αποφυγής, αποφυγής των τραυσμάτων. Σε μία από αυτές τις 50 περιπτώσεις οι αστροναύτες μπήκαν στο Σογιούς, από το Σογιούς μπήκαν στο σωστικό τους ε, όχημα γιατί υπήρχε περίπτωση να υπάρξει σύγκρουση. Αυτό θα ήταν καταστροφή και θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το σταθμό με όλες τις επιπτώσεις ε, και μπορείτε να καταλάβετε ότι θα ήταν και τεράστιο το κόστος. Η επιτήρηση λοιπόν της ε, τροχιάς των θραυσμάτων είναι πολύ σημαντικό. Η οργάνωσή μας συμμετέχει και στους άλλους δύο δομείς. Ο καιρός το διάστημα, άρα είναι ο κίνδυνος από την κοσμική ακτινοβολία, από το πλάσμα, τον ηλιακό ήλιο, τον ηλιακό άνεμο και τα μαγνητικά πεδία. Ξέρετε ότι η κοινωνία μας εξαρτάται όλο και πιο πολύ από ηλεκτρονικό εξοπλισμό στο έδαφος και στο διάστημα. Όταν γίνονται μεγάλα ηλιακά γεγονότα, επεισόδια, πέρυσι είχαμε πολλά τέτοια χρόνια. Όλα αυτά τα, όλα, για παράδειγμα τα δίκτυα, τα ηλεκτρικά δίκτυα, μπορεί να θυγούν. Και αυτό έχει επιπτώσεις για την αέρια κυκλοφορία. Υπάρχουν προβλήματα και για τις συνδέσεις μέσω δορυφόρων. Ε, ε, για παράδειγμα, έμαθα ότι υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας Ιταλίας-Αφγανιστάν λόγω των ηλιακών επεισοδίων. Πρέπει λοιπόν να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Γιατί είναι σημαντικό για, την, για τον ESA αυτά τα ηλιακά επεισόδια ο διαστημικό καιρό δηλαδή, έχουν επιπτώσει στην υποδομή μας. Στις 7 ε, Μαρτίου ένα συγκεκριμένο δορυφόρος παρατήρησε μια μεγάλη ηλιακή ανάφλεξη. Το μελετήσαμε στο, στο κέντρο μας ε, παρατήρησης του διαστημικού ε, καιρού. Μελετήσαμε τι γινόταν, τους δώσαμε στο Ευρωκοντρόλ τη προφορία, αλλά θεωρούσαμε ότι δεν θα είχε μεγάλες επιπτώσεις. Αλλά τρεις από τους δορυφόρους μας εθίγησαν από αυτό το φαινόμενο, το Venus Express, ένα διαστημόπλιο που μελετάει τον, την Αφροδίτη και που μελετάει και τα διαστήματα, ε, τυφλώθηκε το σύστημα ε, πλοήγησής του και χρειάστηκε να το, να το ξαναξεκινήσουμε, να το αναδιαμορφώσουμε. Και το τελευταίο στοιχείο της ε, επιτήρησης του διαστήματος που μας ενδιαφέρει η τρίτη διάσταση είναι τα αντικείμενα που μπορεί να πλησιάσουν τη γη, κομήτες και αστεροειδείς, που δηλαδή ε, περιφέρονται γύρω από τον ήλιο, είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο και μπορεί να προσεγγίσουν τη γη. Παράδειγμα, ένας αστεροειδής που λέγεται απόφυσης ανακαλύφθηκε το 2004 υπάρχει πιθανότητα 2% να ε, προσχρούσει στη γη το 2029. Πρέπει να τον παρατηρούμε λοιπόν. Ξεκινήσαμε το 2008 ένα πρόγραμμα που ονομάσαμε προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για την επιτήρηση του διαστήματος για να μελετήσουμε αυτούς τους τομείς επιτήρηση, ηλιακό κλίμα συμμετέχουν ε, ο Καναδάς η Νορβηγία, η Ελβετία και 13 χώρες μέλη του ESA. Η χρηματοδότησή μας είναι 50 εκατομμύρια ευρώ και θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του 2013. Πριν από ένα μήνα αποφασίσαμε να συνεχιστεί και μετά το πρόγραμμα αυτό για μια δεύτερη περίοδο. Νέα φάση λοιπόν του προγράμματος αυτού, επιτήρηση του διαστήματος, αλλά σε πλήρη συμμόρφωση με αυτά που ανέφερε ο κύριος Μαλακάρνε θα, στο, θα στοχεύσουμε κυρίως ε, το κλίμα και περιορισμένα θα μελετήσουμε, θα έχουμε ε, προγράμματα έρευνας του διαστήματος. Θα συμμετέχουν 14 χώρες μέλη του ESA, θα συμμετέχει και η Νορβηγία και η Ελβετία, είναι οι χώρες μέλη που συμμετείχαν και στα προηγούμενα προγράμματα, αλλά δύο χώρες, η Ισπανία και η Γαλλία που συμμετείχαν, θα αποχωρήσουν θα είναι περίπου 50 εκατομμύρια χρηματοδότηση και της επόμενης περίοδου. Ούτως έχει τώρα η κατάσταση και ευχαριστώ. Ο κύριος Άσμπεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ αγγλικά θα μιλήσω. Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ που μας καλέσατε εδώ πέρα σήμερα και ειδικά την υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης. Θα ήθελα να σας πω πως η υπηρεσία μας ε, έχει εμπλακεί στο σχεδιασμό και στις ε, δραστηριότητες της Κομισιόν όσον αφορά βεβαίως την κατάσταση του διαστήματος και την παρακολούθηση τέτοιων σωματιδίων γιατί υπάρχει μια σημαντική στρατηγική διάσταση στο διάσταμα και στην αντίληψη της ε, κατάστασης και του χώρου. Και όπως είπαν ήδη οι συναδελφοί μου, η οικονομία μας εξαρτάται από το διάστημα, κάθε πολίτης ε, χρησιμοποιεί το διάστημα, είτε μιλάμε για πλοήγηση είτε για επικοινωνίες και τα κράτη στις δραστηριότητές τους, ε, στις σχέσεις τους εξαρτώνται από διαστημικά συστήματα κάθε είδους και αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε πως οι δραστηριότητες ε, και τα γεγονότα στο διάστημα μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τις ε, διεθνείς ε, σχέσεις και την διεθνή σταθερότητα ακόμα αν έχουμε γεγονότα τα οποία είναι σαφή, επιδέχονται παρερμηνία και μπορεί να οδηγήσουν μετά ακόμα και σε κρίσεις. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως ενδιαφέρεται. Επίσης, ως μελλοντικός ιδιοκτήτης διαστημικών υποδομών που είναι κρίσιμες για να σκίσουμε τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνεισφέρουμε στη σταθερότητα και στην ασφάλεια στο διάστημα μελλοντική λοιπόν κατάσταση στο διάστημα. Ε, Η μελλοντική αυτή υπηρεσία παρακολούθησης ε, έχει μια πτυχή και πολιτική και μια πτυχή ασφαλείας. Αυτό αναγνωρίστηκε και σε ένα έγγραφο της ε, Επιτροπής Πολιτικής και Ασφαλείας πριν από ένα έτος που τίτλο είχε «Προώθηση συνεργειών μεταξύ ευρωπαϊκού και στρατιωτικού και πολιτικού επίπεδου, αντίληψη της κατάστασης στο διάστημα και απαιτήσει Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνοψίζει τις ε, απαιτήσει των κρατών μελών στην Πολιτική και Στρατιωτική Επιτροπή. Βεβαίως οι διαστάσεις ασφάλειας είναι πρώτα απ' όλα η ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βεβαίως ε, αφορά παραδείγματο χάρη την παρακολούθηση και προετοιμασία για μη ελεγχόμενες ε, εισόδου ε, δραστηριοτήτων. Είχαμε ένα περιστατικό πριν από λίγου μήνε όπου λόγω της αντίληψη ε, του περιβάλλοντος και της εξάρτησης από τις ΗΠΑ και τη συνεργασία μας με τις ΙΠΑ είχαμε έγκαιρη προειδοποίηση για το περιστατικό αυτό. Βεβαίως υπάρχει μια πτυχή ασφαλείας για την προστασία των ευρωπαϊκών της ευρωπαϊκής υποδομής στο διάστημα. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της ε, ασφάλειας των δεδομένων που απαιτεί ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να χειρίζεται αυτά τα δεδομένα δεδομένης της ευαισθησίας τους και υπάρχει και μια πολιτική πτυχή η οποία, την οποία ανέφερε και ο κύριος Μαλακάρνα η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως θα γνωρίζετε έχει προτείνει έναν διεθνή κώδικα πράση για τις δραστηριότητε στο διάστημα ως ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και διαφάνειας με στόχο πρώτα απ' όλα να συνεισφέρει στην ε, μείωση των ε, διαστημικών ε, σκουπιδιών και συντριπνιών που είναι αυτή τη στιγμή η πιο μεγάλη τεχνική απειλή στις διαστημικές αποστολές Έχει ως στόχο τα μέλη να δεσμευτούν για να αποφύγουν ε, κάθε εχθρική παρεμβολή με τα διαστημικά συστήματα τα συστήματά τους και επίσης υπάρχει η δυνατότητα αμοιβαίας πληροφόρησης για δραστηριότητες, για πρώτερη ειδοποίηση, για εκτοξεύσεις, ε, για συμβάντα όπως προβλήματα με τα διαστημικά αντικείμενα όπως παραδείγματος χάρη διάλυση δορυφόρων η απώλεια ελέγχου δορυφόρων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παρεμβολή με τα διαστημικά συστήματά μας και βεβαίως η παρακολούθηση αυτή του διαστήματος θα συμπληρώσει την πολιτική δήλωση που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση και τα κράτη-μέλη της να γνωρίζει το τι έχουν κάνει τα συμβαλόμενα μέρη που έχουν υπογράψει δηλαδή συνθήκες για το διάστημα όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τέτοιες δεσμεύσεις. Να επανέλθω σε ένα σημείο το οποίο έθιξε ο κύριος Μαλακάρν. Διαβάσατε, κύριε Άσμπεκ, το πρόσφατο έγγραφο σχετικά με τον στρατιωτικό και μη στρατιωτικό συντονισμό. Εξηγήσατε ότι ο εξοπλισμός εδάφους, δηλαδή ραντάρ και άλλα, στρατιωτικής φύσης ε, τα οποία κατέχουν τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να αναπτύξετε λίγο περαιτέρω <clears throat> αυτό το ζήτημα για να μάθουμε πώς, ε, ε, πώς γίνεται η ανταλλαγή, η συνεννόηση, πώς εσείς Κομισιόν λοιπόν κατορθώνετε να συνεργαστείτε με τα κράτη-μέλη, με ορισμένα κράτη-μέλη και με ορισμένα ορισμένες στρατιωτικές δυνάμεις ε, των κρατών μελών. Αυτό είναι μια πληροφορία που θα ήθελα να ακούσω, κύριε Γκάλερ. Ευχαριστώ για αυτά που είπατε. Α, προσοχή γερμανικά. Και για μένα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έμαθα. Για μας πολιτικά είναι σημαντικό να καταλάβουμε την αναγκαιότητα να υπάρχει παρουσία μας σε αυτό το τομέα και να μην είμαστε μόνο καταναλωτές ε, των στοιχείων που μας δίνουν οι Αμερικάνοι φίλοι μας. Η συνεργασία Ευρώπης, είπα και άλλων, που είναι ε, καθοδόν, είναι σημαντική. Η ερώτησή μου αφορά πρώτον τη χρηματοδότηση. Γιατί τάξεις μεγέθους ε, συζητάμε. Αυτό το σύστημα παρακολούθησης. Πόσα χρήματα χρειάζεται. Και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Και μία τεχνική ερώτηση. Το θέμα είναι να δούμε πού είναι τα διάφορα θράψματα για να μπορούμε να έχουμε έγκαιρη προειδοποίηση ή ε, αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο αργότερα να μαζέψουμε όλα αυτά τα σκουπίδια. Ήδη στη γη έχουμε πολλά προβλήματα, στον πολλά προβλήματα και στη γη. Στον ειρηνικό υπάρχουν ε, τεράστια κύματα σκουπιδιών, τα οποία προσπαθούμε να ε, μαζέψουμε και ενδεχομένως να τα αξιοποιήσουμε. Ίσως όμως ε, θα ήταν αποτελεσματικό αν κάποιος θα μπορούσε να τα αξιοποιήσει τεχνικά Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο να έχουμε σύστημα προειδοποιήσεων ούτω ώστε τα διάφορα αντικείμενα που έχουμε στο διάστημα, τα διάφορα σκάφη να αντιδρούν. Ποιες προοπτικές έχουμε να αντιμετωπίσουμε δραστικότερα τα σκουπίδια αυτά. Η Άννα Γκόμες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Φρανζουλιά που ε, αποχωρεί. Θαυμάσια ήταν η εμπειρία μου από την ε, ευσυνειδησία του, την στήριξη που έδωσε στην εργασία μου από τότε που ήμουν την Επιτροπή το 2004. Ευχαριστώ αρμά τις καλύτερες ευχές για τη ζωή μετά το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Καταρχάς, αυτός ο κώδικας δεοντολογίας ε, που θέλει να προωθήσει θέλουν να προωθήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Πώ συνδυάζεται με τι συνθήκε, με τη συνθήκη που υπάρχει από αυτού. Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε αυτή τη συνθήκη για το εξωτερικό διάστημα για το απότερο διάστημα. Και οι άλλοι εμπλεκόμενοι πώς αντέδρασαν σε αυτή την πρωτοβουλία να υπάρξει ένας κώδικας ε, δεοντολογίας. Δηλαδή, ο κύριος Άσμπεκ βεβαίως ανέφερε ότι εξαρτώμεθα από τους Αμερικανούς. Είναι σαφές ότι εξαρτώμεθα απόλυτα. αλλά και άλλοι, όπως η Ρωσία και η Κίνα και ακόμη και η Βραζιλία. Κατανοούν τη σημασία ενός τέτοιου κώδικα, τον αποδέχονται ή αντιδρούν. Και ο Γαλιλαίος πώς μας βοηθάει να αποκτήσουμε περισσότερη ανεξαρτησία στον τομέα αυτό. Τι έχουμε επιτύχει. Και επιπλέον, επιπλέον αυτό το απότερο διάστημα, διάστημα, όλη αυτή η προσπάθεια επιτήρησής του, πώς συναρθρούνται με τα θέματα ασφαλείας ε, επί του εδάφους ή επί και εντός των θαλασσών και σε μεγάλο βάθος μάλιστα, γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Παράδειγμα, αυτή τη βδομάδα στη χώρα μου ένα αεροσκάφος ένα αεροπλάνο που ερχόταν από την Ισπανία θεωρήθηκε ότι αποτελεί κίνδυνο και, και σηκώθηκαν ε, μαχητικά να τον παρακολουθήσουν. Και μετά δεν μας είπαν τίποτα. Τι έγινε αυτό το αεροπλάνο, πού πήγε, προσγειώθηκε πουθενά. Πώς θα μπορούσε το ESA και το Eurocontrol και άλλες, ε, άλλοι οργανισμοί και κυρίως στρατιωτικοί και αμυντικοί, πώς θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να επιλύουμε τέτοια επεισόδια γιατί θα ξανασυμβούν. Τέλος. Τέλος. Υπάρχουν καταστάσεις όπου θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι εάν λειτουργήσουν σωστά θα ενισχύσουν τις δυνατότητες αντίδρασής μας. Γιατί στη χώρα μου άκουσα για παράδειγμα ότι η βάση του Λάζες στις Αζόρες, στη μέση του Ατλαντικού, η, Βα, σεις που βέβαια γεννούν άσχημες αναμνήσεις σε πολλούς γιατί έπαιξαν ρόλο για την επέμβαση στο Ιράκ. Εκεί ανακοινώθηκε η επέμβαση στο Ιράκ. Οι βάσει αυτέ είναι ακόμη σημαντικέ. Τι χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί, αλλά θα αποχωρήσουν. Αυτέ οι βάσει που έχουν όλο αυτόν τον εξοπλισμό που θα μπορούσε να βοηθήσει και για το διάστημα και για το θαλάσσιο χώρο, στρατιωτικό και μη δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Τρία πράγματα θα ήθελα να πω. Πρώτον, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον επικεφαλής της ε, γραμματείας μας που ε, φεύγει. Ένας εξαιρετικός ε, υπάλληλος, σεμνός και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτά που έχετε κάνει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Και τώρα ε, δύο ερωτήσεις που αφορούν το σημερινό μας ε, θέμα. Πρώτον, σε σχέση με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Γκάλερ, ένα ε, συναρπαστικό θέμα. Η είναι πως θα υπάρχουν όλο και περισσότερα σκουπίδια στο διάστημα, δεν θα μειωθούν Οπότε κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε μια κρίσιμη μάζα. Θα είναι πλέον ανεξέλεγκτα. Ο συντονισμός δεν θα επαρκεί και θα οδηγηθούμε σε καταστροφή. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα. Οπότε το ερώτημά μου είναι υπάρχει κάποιος τρόπος να καταστρέψουμε αυτά τα σκουπίδια ή να τα μαζέψουμε ή να τα πάμε σε ένα σημείο. Γίνεται κάτι σχετικά. Κάνουν κάτι οι Αμερικάνοι. Οι υπόλοιποι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει κάτι. Ε, ξέρετε, εμείς ε, στο Κοινοβούλιο Γνωρίζουμε πως έχουμε δυσκολίες στον προπολογισμό, περικοπές, αλλά βεβαίως θα αυξηθεί η χρηματοδότηση της έρευνας και εγώ θεωρώ πως αξίζει να επενδύσουμε σε αυτή την έρευνα. Το δεύτερο ερώτημά μου είναι κάπως πιο προσγειωμένο θα έλεγα. Λάβαμε πληροφορίες από τις ΕΠΑ ότι ένας ε, δορυφόρος μας ε, μπορεί να πληγεί από ένα αντικείμενο. Τι θα συμβεί τότε, πώς μεταδίδονται οι πληροφορίες. Μας ενδιαφέρουν μόνο οι δορυφόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των κρατών μελών. Πώς έχουν τα πράγματα. Γιατί έχουμε δορυφόρου των κρατών μελών που δεν έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται λοιπόν με αυτές τις πληροφορίε γιατί βεβαίω δεν μπορούμε να περιμένουμε να συμβεί ένα ατύχημα. Ο χρόνος είναι... έχει κρίσιμη σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Γκριφόνη Βίντερς, αρχίστε εσεί. Και θα είναι και τα ε, τελικά σας λόγια, επειδή αρχίζουμε με αρίστροφη σειρά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, να αφαιρθώ στα πιο τεχνικά ζητήματα, γιατί υπάρχουν και κάποιες ερωτήσεις που σχετίζονται με την πολιτική διάσταση ή την ε, διάσταση της ασφάλειας. Κάποια πράγματα που θα ήθελα να αναφέρω. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον ζήτημα για, για το τι θα κάνουμε με τα διαστημικά αυτά σκουπίδια. Πράγματι υπάρχει μια πολιτική η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή αυτά τα οποία ανέφεραν οι κύριοι Μαλακάρνε και λοιποί για να τα ταυτοποιήσουμε, να δούμε πού βρίσκονται και Τώρα για το μέλλον είπατε ότι θα γίνουν όλο και περισσότερα. Όχι υποχρεωτικά. Δηλαδή όπως μάθαμε στη γη να ελέγχουμε τα σκουπίδια μας και δεν το μάθαμε αμέσως. Αν θυμάστε πριν από 20 χρόνια πήγαινε κανείς για πικνίκ και τα, τα πέταγε παντού τα σκουπίδια. Τώρα κάνουμε το ίδιο και στο διάστημα. Ε, δηλαδή όταν ε, να αναπτύσσουμε νέα διαστημικά οχήματα, σκεφτόμαστε και το τι θα γίνει στο τέλος του κύκλου ζωής και τι σκοπεύουμε να κάνουμε ε, στο τέλος. Και όταν το εξάζουμε ε, πριν από ένα μήνα στείλαμε ένα πρόγραμμα στα κράτη-μέλη μας ε, το οποίο λέγεται καθαρό διάστημα για το τι θα κάνουμε για να μπορέσει να επανέλθει με τρόπο ασφαλή στην ε, γη ε, χωρίς να δημιουργήσει πρόβλημα και στη γη αλλά ούτε και σε τροχιά. Είναι περίπλοκο το ζήτημα, δαπανηρό, γιατί αναλόγως με το τι υπάρχει ήδη εκεί κάτω, το να το ξαναφέρουμε κάτω σημαίνει άλλη μία αποστολή, αλλά είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε και θα πρέπει στο μέλλον όποτε αναπτύσσουμε διαστημικά οχήματα να έχουν ε, ένα τέλος ζωής με μια ελεγχόμενη επανίσοδο για να μην παράγονται επιπλέον σκουπίδια. Επίσης εξετάζουμε το πώς θα επαναπατρίσουμε κατά κάποιον τρόπο ε, διαστημοπλία τα οποία έχουν βγει εκτό λειτουργία και βέβαια αντιλαμβάνεστε πώ δεν μπορούμε να καταστρέψουμε κάτι τέτοιο γιατί θα δημιουργήσουμε περισσότερα συντρίμια. Οπότε πρέπει να βρεθεί ένα τρόπο συλλογή ή να τα μετακινήσουμε σε μια ασφαλή τροχιά. Αυτέ είναι οι δραστηριότητε τις οποίε εξετάζουμε, ειδικά στα αντικείμενα τα οποία είναι πιο κοντά στη γη, γιατί βεβαίως το, το θέμα σχετίζεται αν... Εντάξει, ο αστεροειδής είναι ένα τεράστιο σκουπίδι αν θέλετε οπότε είναι κάπως παρόμοιο το θέμα αυτά ήθελα να πω τα υπόλοιπα τα αφήσω στους συναδέλφους ευχαριστώ ευχαριστούμε κύριε Σπέκ äh, Ευχαριστώ θα απαντήσω πρώτα στο ερώτημα της κυρίας Γκόμες ε, για τον κώδικα συμπεριφοράς ο κώδικας ε, συμπεριφοράς ε, σε σχέση με το, τις υφιστάμενες συνθήκες ε, για το διάστημα. Υπάρχει ήδη λοιπόν κάποιο δίκαιο για το διάστημα. Ο κώδικας συμπεριφοράς δεν στοχεύει να δημιουργήσει μια νέα νομική βάση. Είναι μια πολιτική δήλωση και τέτοια θα παραμείνει. Δεν θα είναι ε, απαιτητή και νομικά δεσμευτική αλλά ως ε, πολιτική δήλωση θα κινείται μεταξύ των υφιστάμενων συνθήκων και θα είναι αν θέλετε και μία δέσμευση για τήρηση της ε, υφιστάμενης ε, νομικής βάσης. Αλλά σημαντικό είναι πως ο κώδικας αυτός συμπεριφοράς ε, θα αφορά και στρατιωτικές και πολιτικές δραστηριότητες. Και εδώ πέρα έχουμε κάτι το καινούριο. Και εδώ πέρα θεωρούμε πως ε, με την πρωτοβουλία αυτή κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός ανεξαρτήτως από το ότι βεβαίως ε, προσπαθούμε να έχουμε μια κοινή πολιτική, να προτείνουμε μια κοινή πολιτική ε, όσον αφορά την ε, μελλοντική αποφυγή περαιτέρω διαστημικών σκουπιδιών. Γιατί βεβαίως το ζήτημα είναι πως θα πρέπει να εμποδίσουμε την αύξηση των διαστημικών ε, σκουπιδιών με το ρυθμό που είχαν έως τώρα και αυτό είναι ένα βήμα το οποίο δεν θα είναι τόσο απλό. Δηλαδή να οδηγηθούμε σε μία μείωση, αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά αν είναι να περιορίσουμε την αύξηση έχουμε κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός για ε, το διάστημα ως ε, ένα πεδίο δραστηριοποίησής μας. Θέσατε το ερώτημα για την στάση άλλων κρατών. Υπάρχουν τρεις ε, μεγάλες ομάδες, εάν θέλετε. Έχουμε τα κράτη-μέλη που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, αλλά έχουμε και μία σειρά πολύ σημαντικών εταίρων, όπως είπα, η ίδια η κυρία Κλίντον τον Ιανουάριο ρητός ε, ανέφερε και χαιρέτησε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ως μία βάση για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ε, και βεβαίως είμαστε ευγνώμονες αλλά άλλες χώρες όπως η Αυστραλία ή η Ιαπωνία επίσης ε, μας στηρίζουν. Μετά έχουμε τη μεγάλη ομάδα των ε, αδεσμεύτων κρατών που εξέφρασαν ανησυχίες για την ε, συζήτηση του κώδικα αυτού εκτός των Ηνωμένων Εθνών. Αυτός είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα να ε, συζητήσουμε εκτός του ΟΗΕ γιατί θεωρούν πως είναι πιο γρήγορο, πιο πρακτικό και ε, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα γρηγορότερα από ότι μέσω του ΟΗΕ. Βεβαίως τίθεται το ζήτημα μετά πού θα συζητηθεί. Γι' αυτό είναι ρεαλιστική η προσέγγιση μας για να καταλήξουμε γρήγορα σε κάποιο αποτέλεσμα. Μία άλλη πτυχή είναι πως κάποιες αδέσμευτες χώρες εξέφρασαν ε, τον φόβο πως ο κώδικας αυτός ε, αναπτύχθηκε από μια ευρωπαϊκή σκοπιά μια σκοπιά κρατών δηλαδή που ήδη έχουν παρουσία στο διάστημα και ίσως θα περιορίσει αυτές τις χώρες για το μέλλον για την ανάπτυξη και χρήση δηλαδή ε, του διαστήματος από τις χώρες που δεν δραστηριοποιούνται εκεί ακόμα. Γι' αυτό θεωρούμε πως ε, ο στόχος μας είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό ακριβώς θέμε, δηλαδή να διαφυλάξουμε το διάστημα και για το μέλλον και για τις χώρες οι οποίες ακόμα δεν έχουν δραστηριοποιηθεί. Μετά έχουμε χώρες, τη Ρωσία και την Κίνα δηλαδή, που έχουν δικές τους προτάσεις στην ε, διάσκεψη για τον αφοπλισμό στη Γενέβη υπό τον τίτλο «Πρόληψη της ε, τοποθέτησης διαστήματος ε, στο απότερο διάστημα που έχουν ε, το χαρακτήρα μιας συμφωνίας ελέγχου εξοπλισμών και εκεί πέρα εκφράστηκε ο φόβος πως π.χ. ο κώδικας συμπεριφοράς θα μπορούσε να καταστήσει την πρωτοβουλία αυτή χωρίς αντικείμενο. Ε, εμείς θεωρούμε πως ισχύει το αντίθετο πως ε, είναι συμπληρωματικές αυτές οι δύο πρωτοβουλίες και οπωσδήποτε δεν τίθεται ε, ζήτημα αντίφασης με κάποια πρωτοβουλία αφοπλισμού. Αυτά είχα να πω με αυτό το θέμα. Σε αυτά θα μείνω. Ευχαριστώ κύριος Μαλακάρνα. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω το πλαίσιο και να βγάλω κάποια συμπεράσματα. Είδαμε πως ε, το πρόβλημα των ε, θραυσμάτων ε, σχετίζεται με τρία ζητήματα. Να τα αποφύγουμε, να αποφύγουμε την διάδοσή τους και να τα εντοπίσουμε για την κατάργηση, για, όπως είπε και η συνάδελφος, ε, υπάρχουν μελέτες ε, μελλοντολογικές τα έλεγα, φουτουριστικές, αλλά αφορούν ε, τεχνολογίες ιδιαίτερα δαπανηρές που κάποια μέρα θα μας βοηθήσουν στο να καθαρίσουμε κάποιες περιοχές πυκνοκατοικημένες από αυτά τα θράσματα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στείλουμε αποστολές στο κατάλληλο ύψος, αποστολές οι οποίε, όπω είπαμε, θα είναι ιδιαίτερα δαπανηρέ. αλλά χρειάζεται προσπάθεια όχι μόνο οικονομική, αλλά και πολιτική. Να υπάρξει πολιτική βούληση. Πώ να αποφύγουμε την διάδοσή του και γιατί. Ε, ε σε αντιδιαστολή με τα πλαστικά μπουκάλια και τσάντες ε, υπάρχει δυνατότητα να συγκρουστούν αυτά τα αντικείμενα μεταξύ τους και να δημιουργήσουν περαιτέρω φράσματα και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση. Ουδής γνωρίζει το όριο συγκέντρωσης των στρασμάτων. Ε, Γνωρίζουμε μόνο ότι είναι δυνατόν και μια τέτοια είδους αντίδραση θα επηρεάζει σημαντικά την χρήση του διαστήματος ε, ιδιαίτερα σε κάποιες ε, πορείες, σε κάποιες αποστάσεις θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να παγώσουμε τουλάχιστον την σημερινή κατάσταση. Φυσικά χρειάζεται να δούμε τι συμβαίνει και τι θα συμβεί για πολλούς λόγους όπως το θέμα της διαστημικής κατασκοπίας αλλά ας περιοριστούμε μόνο στο θράσματα που βρίσκονται στο διάστημα θέλουμε να γνωρίζουμε πώς έχει η κατάσταση πώς πρέπει να αντιδράσουμε τι χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν πρέπει να έχουμε ένα, μια σαφή εικόνα της κατάστασης το που έχει σημασία είναι να αποκτήσουμε κάποιο σύστημα που θα μας επιτρέπει με τρόπο ανεξάρτητο σχετικά να έχουμε αυτή την ε, πληροφορία. Μια πληροφορία που βρίσκεται ίσω εκτό των δυνατοτήτων και οι ΗΠΑ έχουν ένα σύστημα το οποίο έχει περιορισμού. Βλέπει αντικείμενα από κάποιο μέγεθο και πάνω και, και αντικείμενα κάτω από ορισμένο υψόμετρο οι ΗΠΑ ε, φροντίζουν να ενδυναμώσουν, να το σύστημά τους, ε, αλλά δεν μπορώ να σας πω πόσο θα κοστίσει ένα παρόμοιο σύστημα. Είναι μια πληροφορία, θα έλεγα, απόρριτη. Πρόκειται πάντως για απόρους τους οποίους λίγα κράτη είναι ε, διαθέσιμα να δαπανίσουν. Εξού και η ανάγκη μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυνατότητες ε, και τις ε, υποδομές που έχουμε στην Ευρώπη. Ε, οι οποίες όμως υποδομές βρίσκονται υπό στρατιωτικό έλεγχο. Το Space Council επανειλημμένα τόνισε την σημασία αυτού του είδους συντονισμού υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο μιας κατάλληλης διακυβέρνησης το συγγνώμη που χρησιμοποιώ πότε πότε αγγλικές ε, λέξεις. Η έννοια του governance για να πετύχουμε μια κατάλληλη υπηρεσία για ε, μη στρατιωτικούς σκοπούς είναι ένα ζήτημα πολιτικής φύσης. Γι' αυτό λοιπόν όπως ε, είπε και ο κύριος Νταντζάν, εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάμε με τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες ε, για τον έλεγχο τη χρήση και τη λειτουργία αυτών των ε, υποδομών που όπως είπαμε είναι στρατιωτικές και όταν συζητάμε με στρατιωτικούς ε, και λέμε τον λόγο, τη λέξη governance του σηκώνεται η τρίχα. Τι εννοείται με governance μας λένε. Στο συγγνώμη που κάνω χιούμορ πάνω σε ένα σοβαρό ζήτημα ε, εδώ βρίσκεται το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Συζητάμε και διαπραγματευόμαστε με τι ε, στρατιωτικέ οντότητε, ε, οι βλέπουν με καλό μάτι τη δυνατότητα χρηματοδότηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση για να συντονίσουν αποτελεσματικότερα την ανταλλαγή δεδομένων, χωρί να μπω σε λεπτομέρειε. Η ευαισθησία και η ικανότητα επίλυση του προβλήματος εξαρτάται από τον αριθμό των ραντάρ που είναι διαθέσιμα. Όσο περισσότερο ραντάρ υπάρχουν, τόσο καλύτερα έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο και είναι μεγαλύτερη η δυνατότητα εντοπισμού ε, μικρών αντικειμένων σε μεγάλες αποστάσεις. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ισχυρά ραντάρ, αλλά και θα πρέπει να ε, συζητούν μαζί τους ε, μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν στοιχεία. Και όταν γίνεται ανταλλαγή στοιχείων σε στρατικό επίπεδο, ξέρετε ότι μπαίνει και το θέμα τη ασφάλειας, της εθνική ασφάλειας, άρα η διακυβέρνηση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα έδαφος για την Κομισιόν καινούριο να συζητάμε λοιπόν με στρατιωτικούς, με στρατιωτικές αρχές και να διαπραγματευόμαστε να μελετάμε πώς θα χρηματοδοτήσουμε τις δραστηριότητε του, ώστε να έχουν κάποιες επιπτώσεις στον μη στρατιωτικό τομέα, στον πολιτικό. Αυτό χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά τόσο από μια πλευρά όσο από την άλλη είμαστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι για τις δυσκολίες που υπάρχουν αλλά και για τη σημασία που έχει ο διάλογος. Θα ήθελα να μια παρατήρηση επί των διαστημικών υποδόμων όπως λέει η κυρία Γκόμες και συγκεκριμένα Γκαλιλαίο. Αυξάνει τον Γκαλιλαίο τις δυνατότητές μας, ικανότητές μας σε αυτό το τομέα ή όχι. Η απάντηση εντάχει είναι όχι αυξάνει την ε, ευαλωσιμότητά μας θα έλεγα διότι οι δορυφόροι Γαλιλαίου βρίσκονται εκεί πάνω στο διάστημα και ενδέχεται να πέσουν θύμα θα έλεγα μια σύγκρουση και μια τεχνική λεπτομέρεια οι ε, δορυφόροι ε, για την κυκλοφορία βρίσκονται σε πολύ μεγάλο ύψος, βρίσκονται λοιπόν σε μια ζώνη όπου η πυκνότητα των θραυσμάτων είναι πολύ μικρή. Αλλά όταν ανέρχονται, ανεβαίνουν στο, μετά από την εκτόξευσή τους, όταν πρέπει να φτάσουν στα 200 χιλιόμετρα, περνάνε από περιοχές που υπάρχουν πάρα πολλά θράσματα. Λοιπόν, οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι αυξάνουν την ε, ευαλωσιμότητα της Ευρώπης, ε, άρα την ανάγκη να αποκτήσουμε ένα αυτόνομο σύστημα εντοπισμού. Ναι, από αυτούς τους δορυφόρους, Galileo, δηλαδή GMS, αλλά και ε, δορυφόροι επικοινωνίας, εξαρτώνται οι ικανότητες τις οποίες αναφέρατε, δηλαδή την επιτήρηση της ναυσιπλοείας, την ε, ε, επιτήρηση των αεροσκαφών, αεροσκάφη τα οποία προσγειώνονται έχουν ανάγκη από το GPS, από το Galileo, για να μπορούν να προσγειώνονται ασφαλώς σε αεροδρόμια που έχουν ε, ομίχλη. Ακόμα και αν κάνανε απεργία μια ημέρα σε δορυφόροι τότε θα είχαμε καταστροφές. Όλη αυτή η υποδομή λοιπόν είναι στρατηγικής φύσης τόσο στο στρατηγικό όσο και σε μη στρατιωτικό επίπεδο. Οτιδήποτε εμεί πράττουμε απαιτεί την ε, παρουσία δορυφόρων. αυτό δείχνει ότι είμαστε ευάλωτοι και άρα χρειάζεται ένα σύστημα ε, καθαρισμού, εποπτείας ε, και ελέγχου της διάδοσης Άρα λοιπόν βλέπετε ότι πρόκειται για ένα πλαίσιο ιδιαίτερα περίπλοκο και ευελπιστώ πως ε, θα συνεχίσουμε και τους προσεχείς μήνες ε, θα επανέλθουμε και θα συζητάμε για τις μελλοντικές πρόοδους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ίσως μια ερώτηση που σχετίζεται με αυτά που μόλις αναφέρατε για τις σχέσεις ε, αρκετά καινοτόμες μεταξύ της Επιτροπής και των στρατιωτικών είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει. Ενδιαφέρον. Τι ρόλο παίζει το, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Γιατί νομίζω ότι και εκείνη συμμετέχει στο πρόγραμμα. θα μπορούσε να έχει παραστεί εκπρόσωπός της σήμερα. Τι ρόλο παίζει, πώς αρθρώνεται η συνεργασία σε επαφή με τις ε, ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών, ε, μπορεί να χρηματοδοτήσει ενδεχομένως. Είναι απλώς ως παρατηρητής. Θα απαντήσω αγγλικά ούτως ώστε οι συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας να μπορούν να παρεύουν. Από ό,τι ξέρω δεν συμμετέχουν δεν συμμετέχει αυτός ο οργανισμός στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και κάποιων στρατιωτικών φορέων. Συμμετέχει αυτή η υπηρεσία σε κάποια ερευνητικά προγράμματα. Ήδη έχουμε ορισμένα που καλύπτουν κάποιες πλευρές ε, της επιτήρησης του διαστήματος, το κλίμα στο διάστημα, αντικείμενα στο διάστημα κλπ. Σίγουρα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα έχει τεχνική αλλά και πολιτική αρμοδιότητα, αλλά από ό,τι ξέρω δεν συμμετέχει άμεσα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Επιτροπής και στρατιωτικών φορέων, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερη, ε, καλύτερο συντονισμός των υποδομών του συστήματος επιτήρησης του διαστήματος. Θέλει κανείς από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας να διευκρινίσει? Όχι, ωραία. Ωραία. Α, κύριος Άσμπεκ. η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος στο παρελθόν συμμετείχε ε, στο καθορισμό των αναγκών των χρηστών από την ε, πολιτική αλλά και από την στρατιωτική πλευρά καθορίστηκαν οι προδιαγραφές. Συμμετείχαν λοιπόν στο καθορισμό σε αυτήν την προγενέστερη φάση. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση ενός θέματος για το οποίο οπωσδήποτε θα ξανασυζητήσουμε. Ίσως δεν έχουμε ασχοληθεί επαρκώς ε, με το θέμα αυτό μέχρι τούδε. Δεν ε, θεωρούμε ότι είναι ο κίνδυνος άμεσος. Όλα αυτά συμβαίνουν πολύ ψηλά. Αλλά είναι σαφές ότι οι επιπτώσεις ασφάλειας είναι οπωσδήποτε σημαντικές. Ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας. Θα αξιοποιήσουμε την παρουσία σας και για άλλα θέματα στο μέλλον, για το Γαλιλαίο, οπωσδήποτε. Ο κύριος Γκάλερ, πριν κλείσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Αρμάν για την πολιτική του υπηρεσία. Βγαίνετε τώρα στη σύνταξη και η σταδιοδρομία σας ακολούθησε παράλληλα την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την αύξηση των αρμοδιοτήτων του και βεβαίως άλλαξαν και οι δομές της ε, εργασίας και βέβαια το ζήτημα της ε, Ασφάλειας και της Άμυνας είναι σε μια φάση ανάπτυξης όσον αφορά τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και η πολιτική βούληση βεβαίως υποστηρίχθηκε με τρόπο ικανό από την διοίκηση. Το κάνατε αυτό πάντα και με ανάληψη πρωτοβουλίας, πάντα ήσασταν διαθέσιμος και ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν αυστηρά υπηρεσιακό, σας ενδιέφερε πάντα προσωπικά Γι' αυτό θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία για ό,τι κάνετε από εδώ και μπρος. Και οπωσδήποτε θα σας ε, θυμόμαστε και εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο. Και από μένα λοιπόν καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε με τα λόγια σου διευκρινίσω δύο πράγματα πρακτικής φύσης. Μην εντυπωσιάζεστε που δεν προσφέρουμε κάτι στον αρμό σήμερα, αλλά θα τον καλέσουμε τον Ιανουάριο σε μια συνάντηση, μια μέρα καταλληλότερη, διότι η Πέμπτη δεν είναι και η καλύτερη ημέρα για τους Ευρωβουλευτές. έχουμε ευκαιρία λοιπόν να εορτάσουμε το ζήτημα και με τους συντονιστές και τα μέλη τη Γραμματείας. Θα ε, έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να έχουμε ένα αποχαιρετήριο πάρτι, farewell party όπως λέμε, και να πω ότι συνταξιοδοτήστε, αφιπηρετείτε, αλλά δεν είναι μια ε, σύνταξη, μια στρατιωτικού τύπου. Ξέρω ότι εγκαταλείπεται το θεσμικό μας όργανο μια στιγμή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται και στην καλύτερη φάση. Γνωρίσατε όμως ε, φάσεις και στιγμές πολύ καλύτερες. Δεν πρόκειται για κατάληψη, δεν εγκαταλείπεται το πλοίο όταν ε, δεν τα πάει και πολύ καλά, για να μην Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαι βέβαιος ε, πως στην μελλοντική σας ζωή, εκτός κοινοβουλίου, θα έχετε την ευκαιρία να μας στείλετε κάποια μηνύματα, κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ζωή σας και την προσπάθεια την ευγενή την οποία μέχρι τώρα έχετε καταβάλει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. 36 έτη περίμενα αυτή τη δυνατότητα να λάβω το λόγο και να απευθυνθώ σε ένα κοινοβουλευτικό όργανο. Δράτομαι λοιπόν τις ευκαιρίες. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι πραγματικά με συνεκίνησε ε, η όλη συμπάθεια που ξέφρασαν οι ε, κύριοι κύριοι βουλευτές ε, αυτής της υποεπιτροπής. Είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτή την αντίδραση Εφτά χρόνια είναι επικεφαλής της ε, γραμματείας σας και χάρη στις πρωτοβουλίες σας έζησα στιγμές ε, πραγματικά συνταρακτικές ε, είτε εδώ είτε στις αποστολές που κάναμε στο Τσάντ, στο Κοσμοπέδιο αποστολή στην Παλαιστίνη συγκλονιστικές στιγμές. Είδα λοιπόν την οικοδόμηση αυτής της πολιτικής ε, όταν ξεκίνησε βρισκόμουν στην Επιτροπή Γεωργίας αλλά παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα τεκτενόμενα από τότε την δημιουργία πολιτικο-συνδετικών οργάνων, την πρώτη αποστολή που έγινε στο πλαίσιο της ε, ΚΕΠΑ και Τελευταία είχα και την ευκαιρία να αναλάβω την γραμματεία της υποεπιτροπής σας ε, στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Ήταν μία της περιόδους της πιο συγκλονιστικές ε, και συναρπαστικές. Παρατήρησα λοιπόν πώς ε, οικοδομήθηκε αυτή η πολιτική πετραδάκι-πετραδάκι. Συμβάλαμε κι εμείς στην όλη η προσπάθεια. Να ευχαριστώ του συναδέλφου ε, τη Γραμματεία, που με βοήθησαν σε όλο αυτό το έργο κατά τη διάρκεια των ε, ετών. Ευχαριστώ επίση και του συναδέλφου τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπής του Συμβουλίου και τις υπηρεσίε εξωτερική δράση, δίχως του οποίου το έργο μου θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Οργανώσαμε συνεδριάσει και τους είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων Αυτά. Ολοκληρώνεται λοιπόν στα τωρινή μου 31 Δεκεμβρίου. Διαβεβαιώνω την αναγκόμεση ότι υπάρχει και ζωή μετά το κοινοβούλιο. Απ' έξω θα συνεχίσω φυσικά να παρακολουθώ τι συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποτελεί και τον ε, κοινό μας οίκο. Θα σας σκέφτομαι στις εκλογές του 14 όσοι θα συμμετέχουν τους εύχομαι καλή επιτυχία και επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και ευτυχίες το 2014. 13, συγγνώμη. Merci, euh, merci Armand d'avoir rappelé que nous pourrions nous partir. à... Ευχαριστώ Armand που μας υπενθύμισε ότι εμείς μπορούμε να φύγουμε νωρίτερα. Αυτά είναι οι κίνδυνοι που παρουσιάζει η πολιτική σταδιοδρομία. Θα θέλαμε να σου προσφέρω μια τελευταία συνεδρίαση πιο πολυάριθμη, αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται ε, και στις συζητήσεις αυτές έχει συμβάλει τα μάλα ευχαριστώ για τις δράσεις σου και εκτός της υποεπιτροπής μας. Ε, δεν είναι κατά τύχη, ορισμένοι μπορεί να εκπλήσονται. Όπως είπες, πέρασε από την Επιτροπή Γεωργίας στην Υποεπιτροπή Αμήνας. Ε, ναι, πραγματικά υπάρχει μια ε, συνέπεια. Το λέω, το λέω και έτσι είναι, διότι οι πατέρες ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όταν ξεκίνησαν την ε, αγροτική πολιτική είχαν μια τεράστια πρόκληση να αντιμετωπίσουν και άκουσαν ε, τα ίδια σχόλια και τους προβληματισμούς που έχουμε τώρα στον τομέα της άμυνας. Ε, δεν ήταν αυτονόητο λοιπόν ούτε και τότε. Δεν εφήγησαν τομεί που αφορούν εθνικές, εθνική κυριαρχία, στρατηγική σημασία ζητήματα και είμαι βέβαιο πως υπήρξε πολύ σαρκασμό όταν αυτή η κοινή πολιτική ετέθη σε εφαρμογή. Όταν βλέπουμε λοιπόν το αποτέλεσμα τώρα, την πιστική ασφάλεια, την ε, ε, ε, γεωργική αυτάρκεια, νομίζω ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε συγκλίνει απόλυτα με την δημιουργία τη ε, γεωργική πολιτική. Και νομίζω ότι η πεποίθηση που είχατε τώρα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και για το έργο το οποίο κάνετε εδώ στην Υποεπιτροπή. Ε, χαρακτήρια για την μέχρι τούδε σταδιοδρομία σας, Καλέ εορτέ και ευτυχίες το 2013.